So, dear colleagues, first of all, I would like to welcome the members of the Committee to this joint meeting. Ε, καλημέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω ε, όλους όσους συναδέλφους εδώ και τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΠΕ που παραβρίσκονται, παραβρίσκονται σήμερα μας συνεδρίαση. καθώς εδώ και τον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Μωράς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, θα ήθελα να σας πω στις 14 Νοεμβρίου ο πέμπτος τριμερής διαλόγος έλαβε χώρα στο Στρασβούργο που προβλεπόταν να είναι ο τελευταίος τριμερής διάλογος, αλλά δυστυχώς μας ενημέρωσε εκεί στο Στρασβούργο η Προεδρία ότι δεν είχε κάποια εντολή για να προβεί σε διαπραγμάτευση, ούτε είχε συμβαστικό κείμενο για να προτείνει και κατά συνέπεια η συνάντηση αυτή του τριμερούς διαλόγου ήταν πολύ σύντομη. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι η Προεδρία θα παρουσιάσει ένα συμβαστικό πακέτο για τον επόμενο τριμερή διάλογο που προβλέπεται για τις 13 Δεκεμβρίου και πάλι στο Στρασβούργο. 5η 13 Δεκεμβρίου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Περνάμε τώρα στο ζήτημα που μας αφορά για σήμερα, δηλαδή τους, το κανονισμό για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ένωση. Ε, χαίρομαι το γεγονός ότι και οι δύο επιτροπές μας, η ΛΥΜΠΕ και η ΕΚΟΝ, παραμένουν δεσμευμένες ε, σε αυτή την προσπάθεια της καταπολέμησης ε, του της τρομοκρατίας και του οργανωμένου ο κλίματος. Ε, στις 19 Οκτωβρίου είχαμε κάνει την πρώτη μας κοινή συνεδρίαση για την παρουσίαση της έκθεσης των δύο συνεισηγητών μας, δηλαδή της κυρίας Δελβότη και του κ. Αγγιλά, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή μας λοιπόν κοινή συζήτηση θα εστιάσει στις τροπολογίες που έχουν υποβάλει τα μέλη των δύο επιτροπών μας. Ο στόχος των επιτροπών μας είναι να κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή εκείνων που προβαίνουν σε νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριότητε και των τρομοκρατών όταν εισάγουν ή εξάγουν ρευστά διαθέσιμα από και προς την Άνωση. Μουράς, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας ε, εδώ σήμερα τη Επιτροπή ε, Λίμπε για να συζητήσουμε τον κανονισμό για του ελέγχου αυτών διαθεσίμων. Πρόκειται προφανώ για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Οπότε θα ήθελα να ε, τονίσω και εγώ αυτό που ανέφερε μόλι τώρα ο Πίτες, δηλαδή την ισχυρή δέσμευση των δύο επιτροπών μα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω των ελέγχων των ευστών διαθεσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ένωση. Και δίνω και πάλι λοιπόν το λόγο στον συμπροεδρό μου, ούτως ώστε να δώσουμε τη σειρά το λόγο στους διάφορους ομιλητές μας. Ναι, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουν για 5 λεπτά οι συνεισηγητές, ε, μετά οι σκιώδεις συγητές για 3 λεπτά έκαστος και από εκεί και μετά θα έχουμε και τη διαδικασία catch the eye για οποιοδήποτε συναδέλφους θα θέλουν να πάρουν το λόγο και θα έχουν 2 λεπτά ο καθένας. Άρα λοιπόν δίνω καταρχήν το λόγο στην Μαρή Τελβό, τη μία δηλαδή από τους δύο συνεισηγητές μας, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λάβαμε 263 τροπολογίες. Και προφανώς ε, συμφωνούμε όλοι με το στόχο αυτής της πρότασης, ε, δηλαδή ο κανονισμός για τους ελέγχους δευτερών διαθεσίμων, να ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλήματος ρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είχαμε κάνει και μια ε, συνεδρίαση μεσημεριανού την περασμένη εβδομάδα και νομίζω πως ε, ε, συμφωνήσαμε σε ό,τι αφορά τις τροπολογίε που υποβάλαμε σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ε, μετρητών και κατά πόσο δηλαδή σε αυτόν τον ορισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι προπληρωμένες κάρτες ή όχι. Επίσης υπήρξαν τροπολογίε που υποβλήθηκαν σε ό,τι αφορά τις πληροφορίε οι οποίες θα πρέπει να χορηγούνται σε ό,τι αφορά την δήλωση, σε ό,τι αφορά την διασύνδεση μεταξύ των δικτύων, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε των αρμοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την προσωρινή δέσμευση ε, μετρητών και τη σχετική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ αυτών και των ε, ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης και Κατά συνέπεια, είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν συμβασμό σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη ή όχι των ασυνόδευτων μετρητών σε αυτή τη δήλωση. Η δήλωση δηλαδή προβλέπει αναφορά τόσων των μετρητών που έχει κανείς, ε, των ρευστών διαθεσίμων που έχει κανείς ε, πάνω του, ενώ σε ό,τι αφορά τα ασυνόδευτα ε, διαθέσιμα, παρότι αυτά παρολαμβάνονται στην, στο πεδίο εφαρμογή του οργανισμού, δεν προβλέπεται υποχρεωτική δήλωσή τους. και υπάρχουν λοιπόν κάποια μέλη και των δύο επιτροπών μας τα οποία επιμένουν ότι θα πρέπει πράγματι και αυτά τα συνόδευτα ρευστά διαθέσιμα να δηλώνονται υποχρεωτικά. Εμείς ως συνσηγητές και με τους σκιώδεις συνσηγητές κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και κανείς δεν είναι κατά αυτής της πρότασης, αλλά ε, υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, μια τέτοια διάταξη. Ε, δηλαδή, ποιο θα προβαίνει σε αυτή τη δήλωση, ο αποστολέα, για παράδειγμα, αυτών των ε, διαθεσίμων ο οποίο ενδεχομένω να μην ξέρει ε, από την αρχή ποια θα είναι, ποιο θα είναι το κράτο μέλο εισαγωγή. Οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε είχαν προβλέψει, για παράδειγμα, μια τέτοια υποχρέωση αναφορά αυτών των ασυνόδευτων στον διαθεσίμων στη δήλωση. Και βέβαια οποιοδήποτε είχε κάποια ε, προέβαινε σε αυτή την αποστολή των ωστών διαθεσίμων για παράνομου σκοπούς δεν προέβαινε στη δήλωση. Από εκεί και μετά τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο ο παραλήπτης θα πρέπει να ε, προβαίνει σε αυτήν την ε, δήλωση. Αλλά αυτό τι ε, σήμανε στις ΗΠΑ ότι μόνο εκείνοι των οποίων οι υποβάλλονται σε έλεγχο προέβαιναν σε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή όποιοι κατάφεραν να μην γίνει έλεγχο των αποσκευών του δεν προέβαιναν στην δήλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που εμεί προτείνουμε είναι να περιληφθεί μια ισχυρότατη ρήτρα αναθεώρηση του κανονισμού έτσι ώστε να έχουμε τρία έτη στη διάθεσή μα και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την υποχρεωτική δήλωση την υποχρεωτική αναφορά των ασυνόδευτων ε, στον διαθεσίμων. Οπότε εγώ θα σας πρότεινα να καταλήξουμε σε αυτόν τον συμβιβασμό, σε μια τέτοιου είδου συμφωνία, ότι δηλαδή θα εξετάσουμε τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής μιας τέτοια διάταξη προτού αποφασίσουμε να περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν την ε, δήλωση. Ρίδρα, λοιπόν να θεωρήσεις μετά από τρία χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Αυτά από την πλευρά μου και ο Φερνάντο συνηθίσει ο κύριος Αγγιλάρ θα συνεχίσει σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σημεία τη πρόταση. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνσηγητή της ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Λόπε Αγγιλάρ, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστήθηκα τη συνεργασία με την κυρία Ντελουβό. Λάβαμε 183 τροπολογίες που σχεδόν καλύπτουν όλα τα άρθρα του κανονισμού. Και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμβασμούς που να καλύπτουν όσο να δουν περισσότερες τροπολογίες. Και βεβαίως παραμένουμε ανοιχτοί, ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε. Θα ασχοληθώ με τον συμβασμό 12 και τους επερχόμενους. Ο 12 αφορά το καθήκον της Κομισιόν να αναφέρει ε, τις ε, πληροφορίες που έχει λάβει στις αρμόδιες αρχές. Διάφορες τροπολογίες ε, υποβλήθηκαν για αυτό το λόγο. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας κάποια τεχνικά σημεία, μία αναφορά στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 για την υποχρέωση να δηλώνουν κάποια πράγματα και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κάνουν μία εξοφίσιο δήλωση, ούτως ώστε αυτά τα δεδομένα να είναι προσπελάσιμα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι αυτό ένα μέσο ποινικού δικαίου. Η νομική βάση είναι τελωνιακής φύσεως. Ε, άρθρο 33 της, Ευρω... της Συνθήκης Ευρω... Λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 44. Στο Συμβασμό 14 έχουμε προτείνει να μειώσουμε την περίοδο φύλαξης ούτω ώστε να είμαστε συνεπείς με βάση τις διατάξεις ε, της Europol και τον δονισμο εισοδου εισόδου-εξόδου. Έχουμε δηλαδή προτείνει μία αρχική περίοδο τριών ετών και μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν εγκληματικές δραστηριότητες, που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, η περίοδος θα επεκταθεί σε πέντε χρόνια. Στον ε, Συμβασμό 15 προσπαθούμε να αποφύγουμε το form shopping. Δηλαδή σε περίπτωση ε, που δεν υπάρχει συμμόρφωση θα πρέπει να έχουν ε, αντίστοιχες ποινές στα κράτη-μέλη. Και αυτοί που ξεπλένουν το χρήμα να μην ε, επιλέγουν το πιο επίκες κρατός μέλος. Το άρθρο 14 παραμένουμε στην προσέγγισή μας για τις κατεξουδότηση πράξεις, όχι εφαρμοστικές πράξεις. Ούτω ώστε να έχουμε και εμείς λόγο σε αυτό το θέμα στο Κοινοβουλίο. Στο Συμβασμό 16 προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου για την πρόταση να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα πληροφοριών των τελωνίων, ούτω ώστε να επεκτείνουμε τι πληροφορίε που λαμβάνουμε ε, κατά εφαρμογή αυτού του κανονισμού και έχουμε λάβει διάφορους, ε, υπόψη διάφορου συμβιβασμού που πηγαίνουν προ αυτήν την κατεύθυνση. Στο συμβιβασμό 17, για το άρθρο 18, μιλάμε για την έκθεση που πρέπει να παρουσιαστεί από την Κομισιόν. Ζητάμε την Κομισιόν να αξιολογήσει αν υποχρεωτική δήλωση για το συνοδευόμενα ρευστά, το, το ασυνόδευτο ρευστό θα είναι πιο αποτελεσματική. Το, συζήτησε το είπε αυτό η κυρία Ντελβό. Και η ιδέα είναι, είναι αυτή η προσωρινή ρήτρα που σε περιοδική βάση θα υποβάλει η Κομισιόν, κάθε τρία χρόνια δηλαδή, και μπορεί να αλλάξει αυτό με βάση την εμπειρία. Η ρεαλιστική προσέγγιση που σας εξήγησε η κυρία Ντελβό είναι η βάση για αυτό το συμβιβασμό. Σε αυτό το σημείο του άρθρου 18. Ένα σύντομο σχόλιο για τις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, συμβασμός 18. Ασχολείται με τη θέση για τις ε, προκλειωμένες κάρτες. Έχουμε λάβει ε, διάφορες τροπολογίες που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Συμβασμός 19 οικονομικές μονάδα οικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών και την ανάγκη να υπάρχουν πληροφορίες στις, στα τμήματα αυτά οικονομικών ε, πληροφοριών των άλλων κρατών μελών και ζητάμε από την Κομισιόν να προτείνει μια ευρωπαϊκή μονάδα, ένα ευρωπαϊκό τέτοιο τμήμα οικονομικών πληροφοριών. Και έχουμε λάβει και εδώ υπόψη διάφορες τροπολογίες. στον συμβασμό 20 ασχολούμαστε επίσης με την πρόθεση αποφυγής, με την προσπάθεια να αποφύγουμε το forum shopping σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Συμβασμός 21, και τελειώνω, ε, κοινή διαχείριση του κινδύνου που θα αποφασιστεί από την Κομισιόν μέσω των κατεξιδότηση πράξεων και τέλος. Ένα συμβασμός για την ε, σημασία μιας εκστρατείας αφύπνισης για τους καλόπιστους ε, ταξιδιώτες, επιβάτες. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο νομικό καθεστώς, για το συνοδευόμενο και ασυνόδευτο ρευστό. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων για συμβιβασμούς την Πέμπτη. Θα κάνουμε ένα νέο γύρο για αυτό το θέμα με τους ε, συνεισηγητές και σκιώδεις συγητές. Τώρα, οι βουλευτές να μιλήσουν για λίγο και οι δύο επιτροπές θα συνεδριάσουν από τις 9 και μετά ούτως ή άλλως. Για λίγο ο κάθε ενδιαφερόμενος ευρωβουλευτής. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους ε, εισηγητές και τους συνεισηγητές μάλλον για τη θαυμάσια δουλειά που έκανα μέχρι στιγμής. Όλοι συμφωνούμε για τη σημασία αυτού του κανονισμού και το να έχουμε ένα νέο ορισμό του τι είναι ρευστό. Είναι σημαντικό για να καταλάβουμε επίσης και το νέο μέσο που είναι οι προπληρωμένες κάρτες. Για μένα επίσης τα πολύτιμα μέταλλα είναι πολύ σημαντικό και η πολύτιμη λύθη. Γιατί είναι κομμάτια τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα χρήμα. Επίσης, πολύ γρήγορα, συμφωνώ ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το κείμενο. Η Κομισιόν πρέπει να το αναθεωρήσει, όχι σε πέντε χρόνια, σε τρία χρόνια. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική και ακριβώς γι' αυτό τα τελωνία θα πρέπει να διαβιβάζουν τις ε, πληροφορίες πάρα αυτά. Και επίσης θέλω να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή μονάδα οικονομικών πληροφοριών. Φυσικά θα πρέπει να σεβόμαστε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων και όπως προβλέπει και η απόφαση με το, για το PNR του Καναδά της, του Ιουλίου του 2017. Το θέμα είναι επίσης ποιος έχει ε, πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με τρόπο πολύ λεπτομερή. Για το ασυνόδευτο ρευστό, όλοι συμφωνούν ότι είναι βασικότατο πρόβλημα. Πρέπει να το ρυθμίσουμε. Υπάρχουν υλικέ όμως φυσικές δυσκολίες που μας ε, εμποδίζουν να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό πάρα αυτά, αλλά θέλω να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση όσο πιο αποτελεσματική γίνεται και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα φτιάξουμε ένα καλό κανονισμό και ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του, μέχρι τις αρχές, συγγνώμη, του Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου. Τώρα, για το άλκο κύριο Ματουτσέλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα και για βεβαίω και για όλα αυτά που θα κάνει κατά τι επόμενε εβδομάδε. Οι εργασίε προχωράνε πολύ καλά με κάποια διαφοροποίηση. Υπάρχουν ακόμα θέματα που εκκρεμούν. Ένα θέμα είναι αυτό των προπληρωμένων πιστοτικών κρατών. Αυτέ οι κάρτε χρησιμοποιούνται για πολλά χρήσιμα πράγματα, για ταξίδια παραδείγματο χάρη και έτσι λοιπόν Πρέπει να ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μια μέθοδος που μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς ακριβώς ε, κινείται η ε, χρήση των καρτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Υπάρχουν βέβαια ανώνυμες προκληρωμένε κάρτες και αυτές θα πρέπει να τις εξετάσουμε κατά τις επόμενες συνεδριάσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα που εκκρεμούν. Εμείς έχουμε υπογραμμίσει το θέμα των υπόπτων. Θεωρούμε ότι αυτό το θέμα υποψίες, υποπτή θα πρέπει να ρυθμιστεί και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε κάποιους κανονισμούς έτσι ώστε να ορίζεται ένα ελάχιστο όριο και επίσης και για το απόλυτο όριο των ρευστών διαθεσίμων που μπορεί κανείς να έχει για να μην προκαλέσει υποψίες. 10.000 ευρώ είναι το όριο. Αυτό κατά κάποιον τρόπο μπορεί να ελέγχεται, αλλά στην όλη ε, υπόθεση προβλέπεται η δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε τα ρευστά διαθέσιμα και κάτω από τις 10.000 ε, ε, ευρώ. Εμείς Θεωρούμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί σε σχέση με τους υπόπτους. Ένα άλλο θέμα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες. Τρεις εργάσιμες ημέρες μπορεί να είναι σύντομο χρονικό διάστημα. Ίσως μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Το έχουν προτείνει κάποιοι συνάδελφοι. Ο στόχος του ΕΛΚ είναι με αποτελεσματικό τρόπο να μπορούμε να ελέγχουμε τις κοινή κεφαλαίου για παράνομες πράξεις και θεωρώ ότι για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό κείμενο. Εμείς θέλουμε να σας επισημάνουμε τις τροπολογίες τις οποίες έχει καταθέσει το ΕΛΚ και θεωρώ ότι πράγματι τελικά θα προχωρήσουμε σε αποτελεσματική εργασία, σε καλή δουλειά στο θέμα αυτό. Πρόεδρος, δεν ξέρω, ε, υπάρχει ίσως κάποιος άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο από τη ΛΥΜΠΕ. Όχι, τότε Ίσως ε, κάποιος από την Επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν σκιώδη ηγητές από την ΕΚΟΝ, ο συνάδελφος ε, που ήρθε, ο κύριος Ντεμάζη, α, τον κύριο Ντεμάζη, με συγχωρείτε, άλλοι, δεν ξέρω, υπερβάνσου, στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, συνεισηγητές μας, οι οποίοι με πολύ γοργό βήμα προχώρησαν σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ποιο είναι το διακύβευμα εδώ. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε νέες διαδικασίες για τις ε, διοικητικές αρχές. Είναι, αντίθετα, να δούμε τι κάνουμε με το ρευστό χρήμα το ελεύθερο χρήμα μπορεί να διευκολύνει και το ξέπλυμα και την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και αυτό θέλουμε να το καταπολεμήσουμε με ένα κατόφλι το οποίο είναι αρκετά ψηλό τελικά. Εγώ δεν συνηθίζω να έχω 10.000 ευρώ στην τσέπη μου και δεν ξέρω ποιος το κάνει. Και δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτός που το κάνει. Και μάλιστα, έχω τις υποψίες μου. Αν κάποιος μεταφέρει 10.000 ευρώ σε ρευστό, περίεργο δεν είναι ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη οποιαδήποτε συναλλαγή δεν επιτρέπεται με ρευστό. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε πολλά κράτη-μέλη με ρευστό απαγορεύονται. Γι' αυτό λοιπόν οποιοδήποτε κουβαλάει τόσα λεφτά θα πρέπει να εγείρει υποψίε. Οι δυσκολίε είναι ότι αν δεν υποχρεώσετε να γίνουν δηλώσει, δεν ε, διευκολύνεται και τι κυρώσει. Εάν κοιτάξετε το άρθρο 13 του κανονισμού, λέει, μιλάει για κυρώσεις που συνδέονται με το άρθρο 3 για τα συνοδευόμενα ποσά και το άρθρο 4 για τα ασυνόδευτα ποσά. Για τα ασυνόδευτα ποσά, αυτό ο, αυτός ο μηχανισμός κυρώσεων προβλέπεται για τα κράτη-μέλη. Όπου υπάρχει τέτοια, τέτοιος μηχανισμός, το επιχείρημα ότι σε κάποια κράτη-μέλη θα είναι δυνατόν και σε άλλα κράτη-μέλη θα είναι σχεδόν αδύνατον, αν καταλαβαίνω καλά τις διάφορες παρεμβάσεις, αφήνει αμήχανη. Υπάρχει, υπάρχει ένα ε, μητρό ε, δηλώσεων, ας πούμε, ε, για τα α ποσά, το βάλουμε και για τα β ποσά, ας πούμε. Τώρα, ποιος πρέπει να κάνει τη δήλωση στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνος που στέλνει το χρήμα, έτσι. Σε, ό,τι αφορά τον αποδέχτη τώρα, όποιος λαμβάνει 10.000 ευρώ από το ταχυδρομείο, ή από διάφορους δελιβεράδες. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν ας πούμε, το ταχυδρομείο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να σας δώσει ας πούμε 10.000 σε ρευστό. Δεν μου φαίνεται υπερβολικό να ζητήσουμε το άτομο αυτό να ανοίξει το ίντερνετ του ας πούμε και να πάει να δηλώσει ότι έλαβε αυτά τα 10.000 ευρώ. Ξεπερνάει την κατανόηση ας πούμε αυτό το πράγμα που προτείνεται. Τώρα, η ρήτρα αναθεώρησης είναι ε, αυτή, αυτό το στοιχείο πούμε, που μας καθησυχάζει ως συνομοθέτες, δηλαδή ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε περίπτωση που κάνουμε λάθος. Αν υπάρξουν λάθη, αν υπάρξουν ατέλειες κτλ. Το άρθρο 15 επιτρέπει στην Κομισιόν επίσης, ε, δίνει τη δυνατότητα να, ε, να έχει και εφαρμοστικές πράξεις και για το άρθρο 4 που ισχύουν ήδη. Νομίζω λοιπόν ότι όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν να τροποποιήσουμε το άρθρο 4 υπάρχουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με τρόπο συνεπή. Και υπάρχουν και στις τροπολογίες που κατατέθηκαν και στις τροπολογίες ΓΕΖΕΚ που, δεν είναι εδώ, ε, στις τροπολογίες 167 και 168. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένα συμβιβασμό βάσει, αυτών των δύο τροπολογιών για το θέμα αυτό που σας ε, λέω. Δεν θέλω να δημιουργήσω ένα νέο θάλαμο αερίων. Ε, τις γνωρίζουμε ως λαός, τις ζούμε κάθε μέρα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τι νόημα έχει να κουβαλάει κανείς, ας πούμε, 10.000 ευρώ ε, ή να τη στέλνει με ταχυδρομείο ή με πακέτο εγώ σκέφτομαι απλώς ότι δεν θέλει να ιχνηλατηθούν αυτά τα ποσά, ας πούμε, τα οποία μετά θέλει να τα χρησιμοποιήσει για λαθρεμπόριο, για, για τρομοκρατία κτλ. Και όχι. Και στην πραγματικότητα εμείς ακριβώς αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Επόμενος, ε, ο, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κατσιά, είναι ο κύριος ε, Τσεντεκόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς ε, και είναι δύσκολο να προφέρει το όνομά μου και όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Εγώ είμαι εδώ μόνο για τη συζήτηση και θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτό το θέμα γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς ακριβώς εργάζονται και δουλεύουν οι ποινικοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ αν ήμουν εγκληματία δεν θα πλήρωνα με μετρητά, θα πλήρωνα πλέον με bitcoin. Γιατί πιστεύω ότι το bitcoin είναι το μέλλον όλων αυτών των παράνομων ε, δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, αν θέλει κανείς να πληρώσει ε, για όπλα, για ναρκωτικά, πολλές φορές χρησιμοποιούνται τα διαμάντια. Και αυτό, παραδείγματος χάρη. Θέλω να σας πω ότι την είδα την έκθεση. Η έκθεση είναι πολύ καλή είναι μια έκθεση η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές και όλους τους άλλους που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Εγώ πιστεύω πάντως στο μέλλον ε, πλέον θα συζητάμε για τα bitcoin και για άλλα νομίσματα τα οποία ε, θα υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν Μαρτουτσέλο θέλει να εξανστήσει το λόγο. Δύο λεπτά όμω μόνο, έτσι, γιατί θα πρέπει να τελειώσουμε. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι τα 10.000 ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτήν την έκθεση δεν έχουμε ένα ανώτατο όριο. Για να αρχίσει από εκεί και πέρα να καλλιεργείται μια υποψία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ας πούμε, ε, αν έχουμε κάποιον με 100 ευρώ, ε, αυτό είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να αλλάξουν τα όρια. Ακόμα και αν πολλοί δουλεύουν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. ω εκ τούτου θα πρέπει να βρούμε κάποιον υπάλληλο, τελωνίου, ο οποίος ενδεχομένως επειδή είναι ρατσιστή ή έχει αισθήματα ξενοφοβίας, βλέπει κάποιον ο οποίος για λόγους χρώματος ή για άλλους θρησκευτικού λόγους ενδεχομένως να τον θεωρήσει ύποπτο, ακόμα και αν ο άνθρωπο αυτό έχει μόνο 100 ευρώ επάνω του. Άρα δηλαδή να υπάρχει ένα κατώτατο όριο και εκεί και πάνω να μπορούν να κινούνται οι υποψίες. Το να τα αφήνουμε αυτό έτσι ε, ε, να εκρεμεί, το να μπορεί πλέον να κρίνει μόνος του ο ίδιος ο τελωνικός υπάλληλος ότι θα κάνει όχι ακόμα και κάποια περίπτωση ανθρώπου που διαθέτει 50 ευρώ και να θεωρεί ότι αυτά είναι το αποτέλεσμα ποινικών δράσεων. Ε, αν το κάνω αυτό πλέον δεν είναι κράτος δικαίου. Ε, θέλει κάποιος από του ε, συνσηγητές να ξαναπάρει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρεμβάσει. Δεν νομίζω πως θα καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα σήμερα εδώ. Σε δύο ημέρες θα έχουμε μια συζήτηση και με τους δύο συζητητέ και θα συζητήσουμε το το ζήτημα των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό ή όχι. Πάντως θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι δεν έχει νόημα να θεσπίσουμε ένα κανονισμό ο οποίος δεν θα είναι εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν είμαι υπέρ λοιπόν του να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσο οι προτάσεις που θα κάνουμε είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ε, bitcoins, ε, προφανώς το συζητήσαμε, αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός εδώ ο κανονισμός αποτελεί μόνο ένα τμήμα των εργαλείων που έχουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων κλιματικών δραστηριοτήτων. Ε, το bitcoin δεν θεωρείται δηλαδή νόμισμα και έχουμε άλλα λοιπόν νομοθετήματα εκ των οποίων ένα είναι αυτός ο κανονισμός. Συμπληρωματικά λοιπόν αυτά λειτουργούν προκειμένου να ε, καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Τώρα σε ό,τι αφορά το πώς θα συμπεριφερθεί ένας και μόνο για παράδειγμα τελωνιακός και το πώς εξαρτώνται από αυτόν, νομίζω πως υπάρχει ένα γενικό σύστημα, αν θέλετε, ε, προκειμένου να ε, κριθεί κατά πόσο κανείς είναι ύποπτος ή όχι, ε, σχέτως του αν είναι μεγάλο το ποσό το οποίο έχει ή όχι. Δηλαδή πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται και τέτοιου είδους βέβαια ε, ζητήματα ρυθμίζονται μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Γιατί πάντως και εγώ είμαι της ε, άποψης ότι δεν θα πρέπει όλοι να θεωρούνται εξάντε εκ των προτερών ύποπτοι. Είμαι δηλαδή πεπισμένοι ότι είναι δυνατόν να ακουμπανάει κανείς ε, ρευστά διαθέσιμα πάνω του, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι έχει ε, ε, κάποια κακή πρόθεση. Πάντω σε αυτέ τι περιπτώσει σίγουρα θα πρέπει να έχουν τι δυνατότητε οι τελωνιακοί υπάλληλοι να παρεύουν αν το κρίνουν σκόπιμο και όπω είπαμε θα έχουμε σε δύο μέρε την συνάντηση με του αισιώδει εισηγητέ για να συζητήσουμε περαιτέρω τα αισθήματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμά μα για να μπορέσουμε να περάσουμε το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Νομίζω πω μπορούμε να κλείσουμε την ε, συζήτηση εδώ από την πλευρά τη Επιτροπή ε, ΛΕΒΕ, από την πλευρά του συνσηγητή μα τον κύριο Αγγελάρα ε, και τον, από την πλευρά των μελών της Επιτροπής ευχαριστούμε την Επιτροπή σα για αυτή την πρόσκληση, για αυτή την κοινή συζήτηση σήμερα εδώ και η ψηφοφορία και στι δύο Επιτροπέ ΕΚΟΝ και θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, η Επιτροπή Λίμπε θα συνεδριάσει στην αίθουσα 1α2 στις 9. Και ο κ. Γκουαλτιέρη λέει ότι ε, εδώ στην ίδια αίθουσα